των διαπιστευτηρίων της κυρίας Πύρκο Ρουχόνεν Λένερ και ομόφωνα ε, πρότεινε την έγκριση της εντολής της με ισχύ από τις 27 Απριλίου 2015. Σας προτείνω λοιπόν να εγκρίνετε αυτή την εντολή. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι, ε, εγκρίνεται λοιπόν η εντολή. Έλαβα από την ομάδα... Ε, η ε, ΣΥΑΡ ε, την ε, αίτηση για μια, τη σύσταση, μάλλον μια αναλλαγή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτός ορισμός θα υπάρξει στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί εγκεκριμένη. Μετά από αίτημα λοιπόν, το αίτημα του ομάδα ΕΣΥΑΡ, ο κύριος Σέζα και θα δικαταστήσει τον κύριο Φίτο στην Επιτροπή Περιφερειακή.